Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ξεκινούμε τη συνεδρίασή μας και θα ήθελα καταρχάς να πω ότι έχουμε προσθέσει στην ημερήσια διάταξη την ενημέρωση για τα αποτέλεσματα του τριμερούς διαλόγου σε σχέση με την οδηγία για τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών και το γεωγραφικό αποκλεισμό. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη, με αυτές τις δύο προσθήκες. Εάν ναι, προχωρούμε. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται διαδικτυακά και εύχομαι ένα θερμό καλώς ορίσατε σε όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Υπάρχει η αίτηση για την ηλεκτρονική συνεδρίαση, είναι διαθέσιμη για τα μέλη και τους βοηθούς που επιθυμούν να ε, χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Έγκριση των πρακτικών 24 και 25 Απριλίου του 2017. Τα θεωρώ ότι εγκρίνονται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και γι' αυτό προχωρούμε στην ενημέρωση για τα αποτέλεσματα του τριμερούς διαλόγου μετά την έκθεση της κυρίας Όλγας Σενάλοβα. Πρόκειται για την πρόταση για κανονισμό για τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με το καθήκον της θέσης σε ισχύ της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Όλγα, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον τριμερή αυτόν διάλογο. Ήταν η δεύτερη φορά που γινόταν ε, τέτοιος τεχνικός ε, τριμερής διάλογος σε με περισσότερες από μία συνεδρίες και νομίζω ότι σημειώσαμε αρκετή πρόοδο. Έχει καθορίσει τη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορους τομείς και τώρα περιμένουμε τη γνώμη του Συμβουλίου. Επομένως προχωρούν οι διαπραγματεύσεις και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πολλές και διαφορετικές αναλλακτικές λύσεις. Ορισμένες... Ε, Ορισμένοι τομεί αποτελούν σαφέστατη προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, ισχυρές αρχές και εξουσιοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύει το ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών, ενισχύει το ρόλο των έντιμων επιχειρηματιών και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει περισσότερες δυνατότητες και αρμοδιότητες σε περιπτώσεις παράβασης της κείμενης νομοθεσίας. Θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση και από τα τρία θεσμικά όργανα για να προχωρήσει η νομοθεσία και η εφαρμογή της αν όλοι συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά ενεργητικά όπως το πράττουν μέχρι τώρα, σίγουρα αυτό θα είναι ένα καλό εργαλείο που θα βοηθήσει την καλύτερη εφαρμογή των ε, κανόνων στην εσωτερική αγορά. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για τον επόμενο τρίτο τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, λέει η Πρόεδρος, προχωρούμε στην ενημέρωση για τον επόμενο διάλογο, για τον κανονισμό, για το γεωγραφικό αποκλεισμό και για τη διάκριση με βάση το σημείο εδραίωσης, κατοικίας ή υπηκότητας εντός εσωτερικής αγοράς. Το ρόλο έχει η συγγύτρια. Κυρία Ρούσα, ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, ήταν η πρώτη συνεδρίαση που έγινε και ε, το πνεύμα ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό και στρέφομαι γύρω μου στην αίθουσα, αλλά δεν βλέπω σκιώδεις εισηγητές. Να σας πω ότι και οι σκιώδεις εισηγητές ήταν παρόντες κατά την έναρξη του τριμερούς διαλόγου και παρουσιάσαμε τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πολύ συνεκτικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μια ενιαία και ισχυρή στάση. Νομίζω ότι όλα αυτά λειτουργήσαν πολύ καλά. Βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα και η συζητήση με το Συμβούλιο θα είναι μακροσκελής, πολύ φοβούμε. Να σας πω ποια είναι τα πιο δύσκολα στα οποία πρέπει να επιμείνουμε στο βαθμό του, δυνατού, του δυνατού, όσο περισσότερο μπορούμε. Τέσσερα είναι τα πιο ακαθόδη ζητήματα. Πρώτον, η εφαρμοστέα νομοθεσία. Αυτό το περιμέναμε να είναι δυσεπίλητο ζήτημα, δηλαδή ποιος νόμος εφαρμόζεται όταν οι εταιρείες κατευθύνουν ή δεν κατευθύνουν τις δραστηριότητες τους σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτά πρέπει να περιγραφούν με έναν τρόπο πολύ λεπτομερή, πολύ ε, περιστατωμένο τι σημαίνει κατευθύνω ή διευθύνω τις υπηρεσίες στο άλλο κράτος μέλος. Direct the service. Το Συμβούλιο έχει κάποιο πρόβλημα με τη διατύπωσή μας, αλλά θα βρούμε μια κοινή γραμμή. Ήδη από την πρώτη πολύ σύντομη συνεδρίαση ε, θεώρησα ότι θα βρούμε μια κοινή ε, γραμμή. Δεύτερο θέμα, όταν ο πάροχος περιορίζει τον πολιτή, δεν επιτρέπει στον εμπορευόμενο να πουλήσει διασυνοριακά. Εμείς έχουμε άρρη τον γεωγραφικό αποκλεισμό και μόλις το πράξαμε ή θέλουμε να το πράξουμε. Αυτό είναι πρόβλημα για το Συμβούλιο. Η συμπερίληψη περιεχομένου μη οπτικοακουστικού. Γι' αυτό το θέμα μάλλον είναι ανοιχτό το Συμβούλιο στην πρότασή μας και υπάρχει και η η πρόκληση της ρήτρα αναθεώρησης. Εμείς προτείνουμε την ύπαρξη αναθεώρησης και να υπάρχει αυτό στην νομοθεσία για τη βελτίωση του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Και αυτό αποτελεί ζήτημα πολύ μεγάλης ανησυχίας για το Συμβούλιο. Δηλαδή το ότι θα, ε, το θα συμπεριληφθεί το οπτικοακουστικό κομμάτι στην ε, ρήτρα αναθεώρησης όποτε και αν συμβεί. Ε, σε γενικές γραμμές η συνεδρίαση ήταν πολύ επικοδομητική και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να βρούμε μια λύση σύμφωνοι με αυτά που ψηφίσαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ Ρόζα. Υπάρχουν σχόλια για τον τριμερή διάλογο για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Εάν όχι, περνάμε στην έκθεση της γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό και τις διαδικασίες του 2018 γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Εισηγητή είναι ο Ντάγγελ Ντάντον. Εξετάζουμε τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες. David, έχεις το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σίγουρα όλοι αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι δαπάνες για την εσωτερική αγορά, την ενιαία αγορά. Κάθε ευρώ που δαπανούμε σε αυτό το τομέα φέρνει προστιθέμενη αξία, έχει απτά ωφέλη και επιστροφές στους ε, φορολογούμενους, στους καταναλωτές. Είμαστε όλοι ενωμένοι νομίζω. Δεν μπόρεσα να βάλω τα πάντα ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Προσπαθήσαμε να τις ενσωματώσουμε σε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες που σας έχουμε μοιράσει από την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ το ΕΛΚΑ για την επιπρόσθετη πρόταση στη συμβαστική τροπολογία 3 που προέκυψε από την αρχική τροπολογία 8 του ΕΛΚΑ. Το στηρίζω και στηρίζω τη στήριξη στην καινοτομία. Είναι σαφέστατο το όφελος για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και το Άλντε, τους φιλελεύθερους, για την επικοδομητική τους βοήθεια στις συμβαστικές λύσεις 1 και 2. Μπορώ να στηρίξω τις αναφορές στην βιομηχανία και στα δύο κρατημέλη. Και ως προς τα βασικά της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ, πολλά από τη μελλοντική μας ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα θα εξαρτηθούν από το κατά πώς θα προσαρμοστούμε στην ψηφιακή επανάσταση και αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα του προϋπολογισμού. Ε, οι πολιτικές υπέρ του καταναλωτή, υπέρ των καταναλωτών πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό, το Solvit, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ευρωπαίων Καταναλωτών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ο ενωσιακός τελωνιακός κώδικας είναι πολύ σημαντικός που προβλέπει και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ε, συστημάτων τεχνολογίες και πληροφοριών, το UCC, η απλούστευση ε, και η ενίσχυση των τελωνιακών διαδικασιών είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την καταπολέμηση της αφάτης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης ε, είναι ένας οργανισμός που χρειάζεται στήριξη όπως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και γι' αυτό στηρίζουμε το COSME και το Enterprise Europe Net το Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Επιχειρήν. Πολλές είναι οι προτεραιότητες λοιπόν. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι ως προς τις περισσότερες πρωτοβουλίες. Τελικά να πω ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αξία της επίδειξης δημοσιονομικής ευθύνης. Άρα, άπαξ και δώσουμε προτεραιότητες στις δαπάνες για την εσωτερική αγορά και ε, τις ιεραρχήσουμε, μπορούμε να βρούμε αποταμιεύσεις και εξοικονομήσεις από άλλα σημεία του προϋπολογισμού. Δύσκολο να το πράξουμε με το πλαίσιο το υφιστάμενο, γιατί μπορούμε να προτείνουμε με τη γνωμοδότηση προτεραιότητες για την ενιαία αγορά. ω Επιτροπή αναγνωρίσουμε ότι η ενιαία και εσωτερική αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομεί του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωση που δεν επιφέρουν τόσο μεγάλη προστιθέμενη αξία όσο επιφέρει η κάθε δαπάνη που γίνεται υπέρ τη εσωτερική αγορά. Και αυτό το επιχείρημα πρέπει συνεχώ να το επαναλαμβάνουμε. Σε κάθε περίπτωση ε, υπάρχει γενικότερη έγκριση για τις συμβαστικές τροπολογίες που προτείνουν οι διάφορες πολιτικές ομάδες και ελπίζω η πορεία προς την ψηφοφορία προς τα τέλη Ιουνίου να είναι απρόσκοπτη. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον Αντώνιο από πλευρά ΣΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στα ισπανικά θα τα πω. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Ντάνιελ Ντάλτον, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να συγχαρώ τον Ντάνιελ Ντάλτον για την εξαιρετική δουλειά που κάνει σε αυτή τη γνωμοδότηση και στις συμβαστικές τροπολογίες και θα ήθελα να του ζητήσω να συμπεριληφθεί και το άρθρο 8 στη συμβαστική τροπολογία 3. Ευχαριστώ πολύ που το είπατε και το συμπεριλαμβάνετε, εξαιρετικό Πιστεύω ότι οι βασικές ιδέες που έχουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση είναι μήνυμα προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών, είναι οι πολιτικές ε, ε, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτή που θέλουμε να λάβουν υπόψη για τον προϋπολογισμό του 2018. Μας χαροποιεί όλους που διαπιστώνουμε ότι έχουμε και την εντολή για τα θέματα αυτά του προϋπολογισμού για το 2018 και περιλαμβάνονται οι βασικές πολιτικές γραμμές ε, της Επιτροπής μας, της ΣΥΜΚΟ και αντανακλώνται εδώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω ότι η ενιαία αγορά, όπως κάνω πάντα, ήταν βασικός στόχος ε, οικονομικής συνεργασίας και κυρίως ε, βασικός στόχος ε, για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένω θα πρέπει να υπάρξει επίσης ε, και για αυτές τις επιχειρήσεις ε, ψηφιακή αλλαγή για να μπορέσουμε να έχουμε ε, εκεί ε, ανταγωνιστικότητα, πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές ε, και καινοτομία για τις επιχειρήσεις μας. Πρέπει να επιμείνουμε να υπάρχει κατάλληλος προπολογισμό για το πρόγραμμα Κόσμο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Επιχειρήσεις. Ε, συμφωνούν και πολλοί συνάδελφοι σε αυτό το αίτημα. Τέλος, νομίζω ότι μπορούμε να τονίσουμε ότι το δίκτυο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές θα πρέπει να έχει κατάλληλη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ασκήσουν την αποστολή τους, να εκπαιδεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες για τα δικαιωμάτά του ως καταναλωτέ. Τίποτα άλλο σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο Νικόλα Ντάντι για του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε εκ μέρου τη κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Γκραπίνη δεν μπορεί να παρευρεθεί και επομένω μου ζήτησε να διαβάσω τι σκέψει τη για τι τροπολογίε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του κοιόδης εισηγητέ για την αγαστή συνεργασία. Υπευλήθησαν 16 τροπολογίε. Ε, τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των τροπολογιών των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να υπάρχει κατάλληλος προϋπολογισμός, ο οποίος θα υποστηρίζει τη μετάβαση προς την υλοποίηση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς και μέσω ε, διαδικασιών διεθνοποίησης και ε, νέας εκβιομηχάνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Εδώ επισημαίνω και την ανάγκη να υπάρχει μια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα εξασφαλίζει προστασία των καταναλωτών, αλλά και τη σημασία να υπάρχουν κατάλληλε κατευθυντήριε γραμμέ για μεγαλύτερη ασφάλεια και εποπτεία των προϊόντων, ιδίω στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Ε, τα πρότυπα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα τη εσωτερική αγορά και επομένω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι καταναλωτέ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε αυτή τη διαδικασία προτυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, Επέμεινε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δέουσα σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρχουν και επιχειρηματικά μοντέλα για την κυκλική οικονομία των επιχειρήσεων και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρχουν κατάλληλες γραμμές προπολογισμού που να διευκολύνουν και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες μέσω μελετών της αγοράς, οικονομικών ενισχύσεων και συμμετοχή ε, σε διεθνείς οργανώσεις. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και του στρατηγικού σχεδίου ε, του ΕΦΣΥ για να βελτιώσουμε την ε, ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και προωθούν την έρευνα και την καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ Νικόλα. Για τους σοσιαλιστές δεν βλέπω κάποιον άλλον από τους κοιόδης, επομένως να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Θέλει κάποιος να σχολιάσει. Αν όχι, θα ήθελα απλώ να υπενθυμίσω ότι η αρμόδια επί της ουσίας ε, επιτροπής, ε, ε, η Επιτροπή Προπολογισμών έχει συγγητεί τον κύριο Μούρεσαν. Έχουμε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες συζητώνται. Ήθελα να δώσω την ευκαιρία στο συντάκτη να συνοψίσει στα γρήγορα. Παρακαλώ, Ντάνιελ. Να πω απλώς πολύ γρήγορα ότι συμφωνώ σχεδόν με όλα τα σχόλια που ακούστηκαν από τους συναδέλφους, ιδίω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιστεύω ότι αυτό ε, περιλαμβάνεται στις συμβαστικές τροπολογίες και χαίρομαι που έχουμε ενωμένο μέτωπο. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και προσβλέπω στην ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, ευχαριστώ. Ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ 8 Ιουνίου. και 13 Ιουνίου είναι η προθεσμία για να υποβάλουμε τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο, στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα. Συζήτηση της ε, γνωμοδότησης, του σχεδίου γνωμοδότησης που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Ήτρα. Συντάκτηρα της γνωμοδότησης είναι η κυρία Γκέπχαρτ. Εύελιν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. έχω μια γνωμοδότηση που δεν είναι πολιτικά φιλεγόμενη και την κάνω πολύ πιο ευχάριστα από ότι άλλες γνωμοδοτήσεις, άλλους τομείς. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφου που υπέβαλαν ανθρωπολογίες και που εμπλούτησαν το σχέδιό μου. Έχω κάνει έξι συμβαστικές προτάσεις. Δεν θα έλεγα συμβαστική, αλλά συνο... μια σύνοψη, γιατί δεν υπάρχουν πολλές διαφορές και διαφωνίες. Απλώς συμπερίλαβα και όλες ε, τις απόψεις. Όσον αφορά την πρώτη συμβαστική πρόταση, τονίζουμε ότι πρέπει να αξιοποιήσει την ε, ευκαιρία η Ευρώπη να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μέσω της διεθνικής βιομηχανίας. Στη δεύτερη, ζητάμε από την Επιτροπή να προωθήσει δραστηριότητε που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και που θα οδηγήσει σε ε, ε υψηλά ειδικευμένε θέσει εργασία. Στην Τρίτη, προτείνουμε ότι οι τεχνολογίε διεθνικέ είναι πολύ σημαντικέ για πολιτικέ όπω είναι η αλλαγή του κλίματο, η φυσική πόρη, η μετανάστευση, ο έλεγχο, ο διασυνοριακό και διάφορε άλλε και ότι μπορούν να βοηθήσουν πολύ σε αυτού του τομεί. Στην τέταρτη, Θέλουμε να προωθήσουμε την ε, ευθύνη σε διεθνέ επίπεδο, την ενίσχυση της ευθύνη, να υποστηρίξουμε την χρηματοδότηση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και αυτό είναι κάτι που τονίζουμε στην πέμπτη συμβαστική πρόταση τονίζουμε ότι πρέπει να φροντίσουμε η εμπορικοποίηση των συστημάτων αυτών ότι θα βοηθήσουν ε, τους καταναλωτές και τις εταιρείε και θα πρέπει να δημιουργηθεί για αυτό το λόγο ένα νομικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προστατεύονται τα δεδομένα από παραβιάσεις. και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία νομοθεσία για την αποφυγή της τράπεζας του ανταγωνισμού και επίσης να τονιστεί και ο παράγοντας της ασφάλειας. Θα πρέπει όλα αυτά να ρυθμιστούν και συμφώνησαμε όλοι βέβαια και σε αυτό στην έκτη και τελευταία πρόταση. Στάμε από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τα προγράμματα Έγνος, Καλλιλέο και ε, και Κοπέρνικος να ετοιμάσει την εσωτερική αγορά. Αυτά από την πλευρά μου και πάλι να ευχαριστώ τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες για την πολύ ευχάριστη συνεργασία σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much, ευχαριστώ, Εύελιν. Και τώρα ο λόγος ε, στο ΕΛΚΟ Αντώνιο Λόπες. Thank you, today. So. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή εισηγήτρια, Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το κείμενο. Είναι μια εξαιρετική βάση εργασίας και θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στην Ήτρε ένα καλό προσχέδιο κειμένου. Διαβάζοντάς το, Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να τονίσουμε περισσότερο τα θέματα της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή και γι' αυτό έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Έχουμε προγράμματα διαστημικά επενδύσεων βάσει του ορίζοντα 2020 όπως το Κοπέρνικος και το Έγνος μεταξύ άλλων με στόχο να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, να παρέχονται περισσότερες υπηρεσίες και με μεγαλύτερη ασφάλεια στους καταναλωτές. 230.000 θέσεις εργασίας είναι αυτές που ασχολούνται με τον κλάδο της διαστημικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πλειάδα επιχειρήσεων και η αξία είναι από 46 μέχρι 150 δις ευρώ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις ε, επενδύσεις και τις δαπάνες στον τομέα αυτό βάσει του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2004-2020. Νομίζω ότι θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις μας και θα αποκτήσουν προστιθέμενη αξία. Πρέπει ο ρόλος μας να είναι πρωταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο και να ωφελήσουμε το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε πάρα πολλά ωφέλη από τη διαστημική. Μπορούμε να ε, στηρίξουμε ε, την μετεωρολογία να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ε, εγκαιρότερη και γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση μεταξύ άλλων σε θέματα φυσικών καταστροφών. Ε, είμαστε παγκόσμιος παίκτη και στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης για να, έχει, να κατακτήσει το διάστημα και να ε, ενισχύσει την ασφάλεια αυτού, προωθώντας πάντοτε τη διεθνή συνεργασία. Τα δεδομένα και οι υπηρεσίες που προκύπτουν από τα διαστημικά συστήματα συμβάλλουν στη δημόσια πολιτική σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα στη γεωργία, στον έλεγχο των πληθυσμών, στην ανείχνευση ε, των πετρελαιοκυλιδών όταν είναι όλα αυτά αποτελεσματικά μπορούμε να προωθήσουμε την ενίσχυση των υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων και να ενισχύσουμε τις διάφορες ηλεκτρονικές ή διαδικτυακές εφαρμογές. Και γι' αυτό θα πρέπει τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία συνδέονται τα δεδομένα να είναι διαλειτουργικά. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να καταστούν σαφή στην γνωμοδότηση αλλά και η προστασία του καταναλωτή. Όταν οι συμβαστικές τροπολογίες ε, υποβάλλονται θα ήθελα η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 να περιλαμβάνει περισσότερα από την τροπολογία υπαριθμών 2 που έχω εγώ υποφάλει. Αν αυτό είναι δυνατόν να σας πω ότι για μας το διάστημα δεν είναι κόστος αλλά είναι επένδυση με πολλά και σημαντικά ωφέλη και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Με ανησυχεί κάπως η συμβιβαστική τροπολογία 5 αλλά το γραφείο μου θα υποβάλει σχετική πρόταση πριν λήξει η προθεσμία αύριο. Ευχαριστώ. Ο Ντανιέλ Ντάλτον από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Φυσικά και υπάρχει συνένεση σε αυτό το θέμα και συμφωνούμε όλοι για τις ωφέλειες που μπορεί να έχει στην ε, καινοτομία και συγκεκριμένοι τομείς βιομηχανίας που μπορούν να φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα στις επενδύσεις. Θέλουμε ε, να εξασφαλιστεί ένα ψηλότερο προπολογισμό για τη διαστημική έρευνα. Όμω, θεωρώ και θα προτείνουμε μια τροπολογία εδώ ως ε, παράταξη. Θέλουμε την διαμεσονική ουδετερότητα στην διαστημική στρατηγική και αν όχι αναγνωρίζοντα αυτά που είπαμε για τον προπολογισμό, να ζητήσουμε αύξηση επενδύσεων σε κάποιου τομεί. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι παράλληλα, να είμαστε σίγουροι ότι θα μειώσουμε ε, τον προπολογισμό σε άλλε περιοχέ, γιατί μπορεί να είναι μαύρη τρύπα, όπω καταλαβαίνετε, η διαστημική έρευνα. Γιατί είναι απεριόριστη η δυνατότητα, ε, δυνατότητε έρευνα και γι' αυτό είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Επίσης το ECR πρότεινε μια ακόμα τροπολογία για να ενθαρρύνει την ε, δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Όλοι συμφωνούμε στα θετικά αποτελέσματα ε, των επενδύσεων και για την οικονομία και θα πρέπει να επιφελθούμε στο μέγιστο φυσικά πέρα από όλα αυτά Αυτά θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η συγγήτρια και θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Όπως είπατε και στην αρχή είναι πολύ ευχάριστη ε, η εργασία γιατί δεν έχετε να κάνετε με ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα. Ευχαριστώ για το άλλο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο προηγούμενο Σκιώδης τα είπε καλά. Υποστηρίζουμε αυτά που υπόθηκα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράξει τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, για τις μικρές, επιχειρήσεις, να υπάρξει μια σταθερή συνεργασία. Όλα αυτά είναι προφανή. Τώρα, κοιτώντα τι τροπολογίε, βλέπω μια ανάγκη να τονίσουμε την σημασία μια θετική γνωμοδότηση με εστίαση στα ακόλουθα. ένα πιο φιλόδοξο κείμενο κάνει λόγο για τις στιμικές ε, στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ε, ανάπτυξη. Αναφέρομαι στην τροπολογία 3. Θα πρέπει επίση να υπάρχει παρατήρηση των ε, διεθνικών δεδομένων μέσα από πλατφόρμες ώστε να προκύψει μια εσωτερική αγορά για διεθνικά προϊόντα Υπάρχει μεγάλο δυναμικό και εκεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είναι καλό να το γνωρίζουμε και αυτό. Και κατά τρίτον, όσον αφορά την αθεώρηση του κώδικα για τις τηλεπικοινωνίες και τις εσωτερικές υποθέσεις της εσωτερικής αγοράς, θα ήταν καλό να ενισχύσουμε τη διατύπωση για την δορυφορική τεχνολογία που μπορεί να αποβεί πολύ αποδοτική για τη δημιουργία δικτύων σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα πρέπει να κάνουμε χρήση του δυναμικού που υπάρχει σε αυτή τη βιομηχανία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι τα σημαντικά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλος και όλος που θέλει να πάρει το όλο η Τζούλια Ρέντα. πάμε στην ώρα φτάστε για να μιλήσετε για τους πρασίνους. Take your time. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Κέπχαρντ για τις συμβαστικές προτάσεις. Με πολλές θα συμφωνήσω. γιατί λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις μας. Υπάρχουν δύο επιπλέον τροπολογίες που παρουσιάσαμε, που βάλαμε προστιθέμενες παράγραφοι που δεν καλύπτονται από τις συμβαστικές, όπου θα θέλαμε να ρωτήσουμε την στήριξη της συγκεκριτήρας και των άλλων παρατάξεων, γιατί τα θεωρούμε σημαντικά στοιχεία για τη διαστημική στρατηγική. Το πρώτο είναι η τροπολογία 16 και η δεύτερη είναι 23 για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους της ε, στρατηγικής, θα πρέπει πρώτα να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών και προϊόντων οικολογικού design. Αυτό είναι σύμφωνο με αυτό που ήδη κάνει η ESA, ο ESA και συμπεριλαμβάνει τέτοια πρότυπα στο Clean Space ε, Initiative, στην πρωτοβουλία για το καθαρό διάστημα. Αυτή είναι μια βέλτιση πρακτική και θα πρέπει να το προβάλλουμε αυτό. Γι' αυτό προτείνουμε για την ε, τροπολογία 16 και στην 23 ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν την ε, ευρεία χρήση των προγραμμάτων ε, συστημάτων κρυπτογράφησης για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών και την αθεκτικότητα των υποδομών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους φορολογούμενους που χρηματοδοτούν αυτές τις τεχνολογίες θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα χρήματα δεν επενδύονται σε ευάλωτες δομές αλλά σε υποδομές που χρησιμοποιούν ισχυρές τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ότι οι μελλοντικές επενδύσεις θα είναι ανθεκτικές. Ελπίζουμε λοιπόν όλοι να συμφωνήσουμε ότι η αρχή της ε, προφύλαξης, της πρόληψης θα πρέπει να τηρηθεί όταν ζητάμε και περισσότερη χρηματοδότηση ειδικά για αυτόν τον τομέα. Οπότε με τις και με αυτές τις δύο τροπολογίες θα είμαστε μια χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, εισηγήτρια. Ευχαριστώ Τζούλη. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα θέλει να πάρει το λόγο. Τότε λοιπόν σας ε, θυμίσω ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 8 Ιουνίου και στην Ήτρε θα γίνει η ψηφορία στην 21η Ιουνίου και τώρα πάλι ο λόγος στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω, είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους που θέλουν να εργαστούμε περαιτέρω επί του θέματος όσον αφορά την τροπολογία 2 και τις επενδύσεις. Φυσικά και θα πρέπει να το δούμε με θετικό βλέμμα, αλλά θα ήθελα να το δω και γραπτό. Θα ήθελα να μου περισσότερο και γραπτά. Ο συνάδελφος από το ΑΕΛΚ, λυπάμαι δεν θυμάμαι, να μου υποβάλλετε γραπτά τις προτάσεις σας για να μπορώ να τις δω και να τις συμπεριλάβω Καταλαβαίνετε γερμανικά, σας βλέπω μια χαρά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις για την 2 και για την 5. Ζητάω να μου τις υποβάλλετε γραπτά και είμαι σίγουρη ότι θα βρω μια πολύ καλή λύση. Είμαι υπέρ των επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα όταν είναι απαραίτητες. Αν μου τα επεξηγήσετε επομένω ε, περαιτέρω θα μπορούσα να βοηθήσω. Τώρα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και την έρευνα ε, της ε, τεχνολογίας κρυπτογράφηση και, και όλα αυτά που αναφέρατε και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά. Θα σας δώσω και σύντομα και το voting list για να δείτε πώς θα φανούν ε, οι προτάσεις των τροπολογιών. Αλλά κύριε Ρέντα, θα ήθελα και από εσά να μου δώσετε τι ε, προτάσεις ε, γράφου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Εβελίν. Και εδώ ολοκληρώνουμε το διάλογο για τη διαστημική, διαστημική στρατηγική. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε στις 4 ακριβώς για την ψηφοφορία. ευχαριστώ πολύ.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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

τον Τζόνα Καμπύλα.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

Any socialist wants to give me the voting list? Μήπως κάποιος σοσιαλιστής θέλει, χρειάζεται τον κατάλογο ψηφοφοριών ή μπορεί να μου τον δώσει. Salut, ça va bien Bien toi, ça va Ça va, ça va. Bon. On peut t'asseoir ici Non, je vais mettre... Okay. Καλώς, συνάδελφοι, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε όλοι. Έχετε όλοι τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εσείς δεν τις έχετε. Καλώς θα σας περιμένουμε. Έρχεται, θα σας τη φέρουν. Ίσως διανατάσεως χειρός. Όχι, έρχονται. Okay, Okay, Καλώς. Ξεκινούμε με την ψηφοφορία για τη διασυνοριακή μεταφορά δεμάτων. πια Όρσεν, η συγκήτρια. Είναι εδώ. Καλώς. Γεια σας, θέλετε το λόγο. Όχι, ωραία. Τέλεια. Προχωρούμε στη ψηφοφορία. Τροπολογία 47. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να την ελέγξουμε την 130 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. 131 και 132 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 18α. Τη βρήκατε. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19α υπέρ, κατά, Άποχες εγκρίνεται. 228, 229 είναι ταυτόσημες Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 20. Την ψηφίζουμε ομαδικά μαζί με τη συμβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 268 τροπολογία. 273. Ομαδικά τις ψηφίζουμε γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Να το ελέγξουμε ε, ηλεκτρονικά. Επαληθεύουμε. Από τη 268 μέχρι τη 273 σε μπλοκ τις ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. Καλό, συγγνώμη. 2.84. Όχι, 2.85. Συγγνώμη, 2.85 ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, καταπίπτει. καταπίπτει διότι η 268 εγκρίνεται. Άρα 285 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Ομαδικά με την συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τη 46. Πέρας. Εγκρίνεται. 48. Προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 1. Στις αιτιολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία θέλετε να το ελέγξουμε κανείς δεν το ζήτησε αλλά μπορούμε να το ελέγξουμε ψηφίζουμε την 53 Ψηφίστε συνάδελφοι, ψηφίστε παρακαλώ. Καλώς πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία... Όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 55 υπέρ. Όχι, 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 55. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 καταπίπτει και γι' αυτό πάμε στην 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές το ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 67. Εγκρίνεται. 18 υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά άποχες το ελέγχουμε, το επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 76 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική υπαριθμών 7 όχι, δεν χρειάζεται Πάμε στην τροπολογία 83. Υπέρ κατά αποχές συμβιβαστικές. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 83 ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 καταπίπτει. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 ταυτόσημη με την 103 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε, να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την 104 πέρας απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 και 106 ταυτόσημες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 καταπίτη 108 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 108 Πέρασε εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Δεν έχει ψηφιστεί, δεν ψηφίζεται και πάμε στην 114. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική έναρξη ψηφοφορίας εγκρίνεται 28 ψήφοι υπέρ 6 κατά 2 αποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα, συνάδελφοι, περνάμε στην έκθεση για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρμογή του κανονισμού 1025 του 2012. Η συγγήτρια, η Μαρλέν Μίτσι. Θέλετε να πείτε κάτι? Έχετε το λόγο, κύριε Μίτσι. Θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερως ε, τους και οδησηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα ε, και φυσικά και τους ε, συμβούλους. Και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Περνάμε στην ψηφοφορία, συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 της Στραν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 11 της Ήτρε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 της Ήτρε, υπέρ, α, θεωρείται ότι εγκρίνεται. Συγγνώμη. Τροπολογία 6 της Τραν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της τραν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, ήτρε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 58, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Επαλήθευση της 59, πέρασε της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 19 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία 8 της τραν. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε παλήθευση. Της 63. Επαλήθευση της 63. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Και πάμε τώρα συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 36 Τη Ήτρε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της Τραν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην Ήτρε 20. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τραν 11 Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. συγγνώμη, τροπολογία 3 τραν. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Υπέρ, κατά, απόχέ, επαλήθευση για την 76. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 78. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 17, υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Ήτρε 27, υπέρ, κατά, απόχέ, επαλήθευση της Ήτρε 27. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Ήτρε 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση της 97. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Συνάδελφοι, είναι πολύ κοντά η ψηφοφορία. Σας παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε επαλήθευση για όλες. 17 υπέρ, 17 κατά, καταπίπτει. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Κάποιοι ψήφισαν και υπέρ και κατά. Συνάδελφοι, αποφασίστε. Επαλήθευση λοιπόν, εκεί δεν έχετε δικαίωμα επιλογή. Επαλήθευση της 99. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. 19 υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία 100 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ, υπέρ, 103, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Σας παρακαλώ δείξτε τι ψηφίζετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 113, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τραν 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 118, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 τραν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση της 125. πέρα ψηφοφορία. ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 126 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία. Α, συγγνώμη. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. Τροπολογία 129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 138 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 150. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 156 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές εκθέσεις. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά Σας παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Επαλήθευση επευθείας για να τελειώνουμε. Τροπολογία 1. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ο Νικόλα θέλει επαλήθευση. Εντάξει. Πέρας τη Εγκρίνεται. Σωστά. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Επαλήθευση της 15. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 17. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο. Διαφορά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία α, επαλήθευση της 23, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία α τραν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε τελική ψήφος ηλεκτρονικά, συνάδελφοι. Εγκρίνεται 34 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ολοκληρώνεται λοιπόν η ψηφοφορία για τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του κανονισμού 1022. 1025. Προχωράμε στην επόμενη ψηφοφορία. Σας παρακαλώ να σκόνετε τα χέρια σας. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα προϊόντα, ωφέλη για τους καταναλωτές και τις εταιρείες. Και ο Πασκάλ Τζιγόν, ο εισηγητής, ήθελε να πάρει το λόγο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57. Υπέρ, κατά, αποχές, απόρριπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται 19 προς 16. Συνεχίζουμε στην 125 η οποία εκπίπτει. Στην 127 λοιπόν υπέρ κατά αποχές την ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 127 πέρας. Απορρίπτεται Συμβαστική 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές την απαλληφεύουμε. πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται κατά μία ψήφο. 144 και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 18 προς 17. Εκπίπτει 145, πάμε στη συμβαστική 13, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 151 αποσύρεται. Συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 172. Υπέρ, κατά, αποχές, απόρριπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 17α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 205. Άρχεται η ψηφοφορία. On 205 and the vote is... Πέρας ψηφοφορίας. 18 προς 17. Απορρίπτεται. 206. 207 άρχεται η ψηφοφορία. Έχω και όπως πάντα και απορρίπτεται 20 προς 15. Προχωράμε στην 209 και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 224 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και Απόρριψε 17 προς 17. Άρχεται η ψηφοφορία για την 225. Πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται 17 προς 17. Προχωράμε στην NV3. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σε μπλοκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV6 εγκρίνεται NV8 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε NV8 ψηφίζουμε και εγκρίνεται 19 προς 15 NV9 εκπίπτει και πάμε στην 10 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV12 εκπίπτει πάμε στην 15 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV16 NV16 εγκρίνεται Μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδικά από το 17 μέχρι την 26 για την ΕΝΒΗ. Συμφωνείτε 17 τότε υπέρ. Όχι σε μπλοκ. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. ΕΝΒΗ 19. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία και απορρίπτεται. NV20. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία και απορρίπτεται πάλι 17 προς 17. NV21. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται και αυτή με μικρή διαφορά. 23. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. NV25. Άρχεται η ψηφοφορια πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται κατά μία ψήφο NV26. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. NV27 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. NV31 υπέρ κατά τα αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. Πάμε στην 39. Πέρα στις ψηφοφορίες και απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Μπορούμε, συνάδελφοι, την 40 μέχρι 49 να ψηφίσουμε συνολικά. Τότε μία, μία η 40 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται 15 προς 15, έμβη 41 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία και εγκρίνεται. NV46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV47 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. NV47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV48 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Πάμε στα... On block 18 to 22. Σε τελογικές θέσεις. Μία-μία. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά απορρίπτεται πάμε στο προημείο recitals, αιτιολογικές σκέψεις. And it is adopted. Εγκρίνεται η 4. Αιτιολογική σκέψη 5. εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 6. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. 7. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Αιτιολογική σκέψη 8. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 9. Ναι. Άρχεται ψηφοφορία. Εκπίπτει. NVB. Υπέρ. Κα... Εκπίπτει και αυτή. Πάμε στην 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 12 πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται τροπολογία 13 εκπίπτει και η 14 και η 15 εκπίπτει η 15 εγκρίνεται NVA, άρχεται ψηφοφορία και πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. NVJ, άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. NVL, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται κατά μία ψήφο. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 εγκρίνεται 30 εγκρίνεται 31 άρχεται η ψηφοφορία και απορρίπτεται 32 ψηφίζουμε. Πέρας. Και απόρριπτεται. 17 προς 17. Τροπολογία 33. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34. Άρχεται ψηφοφορία. πέρα και απορρίπτεται κατά μία. 35. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Πέρα ψηφοφορία απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ αποχές απορρίπτεται 39 άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται 40 ψηφίζουμε πέρας και απορρίπτεται τροπολογία 41 ελέγχουμε πέρα ψηφοφορία και απορρίπτεται κατά μία ψήφο 42. Ψηφίζουμε για τη 42, πέρα ψηφοφορία και εγκρίνεται τροπολογία 43, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και εγκρίνεται NVC. NVC ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. NVD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NVE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NVF. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. NVG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NVH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NVI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NVK άρχη ψηφοφορία Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Πάμε στην NVM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NVN ψηφίζουμε και εγκρίνεται NVO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MVP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NVQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική ψήφος πέρας ψηφοφορίας 34 προς 0 μία αποχή συγχαρητήρια στην ε, συγγήτρια, στην συγγητή ολοκληρώνουμε για σήμερα την ψηφοφορία. Σας παρακαλούμε να μείνετε μαζί μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Πάμε στο επόμενο σημείο, στην ημερησία διάταξη. Και όσοι αποχωρείτε από την αίθουσα, παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως. Ζήτησα από τους συντονιστές να παραμείνουν.